Uh, well, uh, Καλή μέρα. Είμαστε στο δεύτερο πρωινό της συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Υπάρχουν και διάφοροι που μας παρακολουθούν ε, από το διαδίκτυο, οπότε γι' αυτό ξεκινάμε. Στην Κρακοβία είχαμε ένα φόρουμ το Σαββατοκύριακο για την ε, εσωτερική αγορά και είδαμε ότι εκεί πέρα ισχύει στα πανεπιστήμια το τέταρτο. Δηλαδή ότι ξεκινούν λίγο αργότερα. Εμείς ε, όμως ξεκινάμε στην ώρα μας γιατί έχουμε εδώ τον εισηγητή μας για μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση που έχει να κάνει με το Γραφείο Εναρμόνισης στην εσωτερική αγορά για τα εμπορικά σήματα και σχέδια. Υπάρχει εδώ πέρα μια πολύ σημαντική πρόταση για την Επιτροπή μας. Έχουμε γνωμοδότηση εμείς για την Νομική Επιτροπή. Ο Άνταμ Μπίλεν από τη ΣΥΑΡ, ο συναδελφός μου, είναι εισηγητής για την πρόταση αυτή και ελπίζω ότι το ΕΠΠ θα μας τιμήσει με τους σκιώδες εισηγητές, την κυρία Μπάστο στο ΕΛΚ και οι υπόλοιποι εδώ, ο κύριος Κρότσμαν είναι ήδη εδώ και περιμένουμε να δούμε αν θα έρθουν και άλλοι. Αλλά έχουμε εδώ βλέπω και μια δυνατή ομάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κυρία Μπέσεβα και τον κύριο Φόρτς από την ε, ομάδα, από τη μονάδα μάλλον για την ε, παραποίηση και την πειρατεία και την κυρία Φανεγκρίν που είναι από το Γραφείο Αναρμόνησης για την εσωτερική αγορά. Καλώς ήρθατε. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν δίνω το λόγο στον εισηγητή για να μας παρουσιάσει τις ιδέες του όσον αφορά αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Κύριε Μπίλεν, ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή είναι μια γνωμοδότηση που ετοιμάζουμε, όπως είπε πολύ σωστά και ο Πρόεδρός μας. Και έχει να κάνει με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εναρμόνιση της τυποποίησης στο Ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πρόκειται για θέματα που έχουν να κάνουν με τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και έχουν να κάνουν και με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την παραποίηση και την πειρατή. Όλα αυτά αναφέρονται στον τίτλο και στην, ε, στον τίτλο της νομοδότησης λίγο πολύ. Επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή είναι νομική επιτροπή το χρονοδιάγραμμα πρέπει να επιταχυνθεί, πρέπει να βιαστούμε. Και εμείς και εκείνοι στην αρχή έπρεπε κατά την Πολωνική Προεδρία να εγκριθεί η έκθεση αυτή, ο κανονισμός αυτός. Δεν ξέρω όμως αν θα τα καταφέρουμε μέχρι το Δεκέμβριο. Κατά πάσα πιθανότητα θα αναβληθεί η έγκριση. Η Επιτροπή μας όμως αποφάσισε να μείνουμε στο αρχικό χρονοδιάγραμμα. Το έγγραφο αυτό έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραπίσης και Πειρατείας που ιδρύθηκε ε, από πρωτοβουλία του Συμβουλίου και της Επιτροπής και στην αρχή ε, δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει το κίνδυνο ε, εμπορίο με παραπημένα προϊόντα και την πειρατεία επίσης στο εμπόριο και εξελίχθηκε σε κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για τη συγκέντρωση και παρακολούθηση και διαβίβαση πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με την προσβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Και αυτό που πρέπει εδώ να τονίσουμε είναι ότι είτε από την αρχή το Συμβούλιο και η Επιτροπή επέκτηναν την εντολή καταρχήν βάσει απόφασης της 1ης Μαρτίου πέρυσι σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά και το παρατήριο ξεκίνησε να αναλαμβάνει και άλλες αρμοδιότητες και να υιοθετεί προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας. Το Κοινοβούλιο άρχισε να συγκεντρώνει και επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά ε, προϊόντα πλαστά. Κατά συνέπεια, μετά την γνωμοδότηση που είχαμε από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, συστάθηκε το εμπορίο αποτελεί, το παρατηρητήριο να αποτελεί και το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Επιτροπή και τις εξωτερικές μας επαφές όσον αφορά την διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Αυτά λοιπόν έκανε το παρατηρητήριο τα δύο αυτά τα τελευταία χρόνια. Επέκτηνε δηλαδή τις δραστηριότητε του κατά πολύ. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει και περισσότερους πόρους οικονομικούς ή προσωπικού έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο προτείνουν τώρα να ανατεθούν αυτές οι επιπλέον αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Αλικάντε. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία για το ότι η Επιτροπή μας ε, πρέπει να ετοιμάσει γνωμοδότηση γιατί ο κανονισμός σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζει και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του καταναλωτή. Σας υπενθυμίζω δε ότι πολλά παραπημένα προϊόντα είναι επικίνδυνα και απειλούν ακόμα και την υγεία. Τα φάρμακα για παράδειγμα, αλλά και τα παιχνίδια οι ηλεκτρικές συσκευές. Συνεπώς, είναι θέμα δικαιωμάτων του καταναλωτή και θέμα υγείας. Έχω υποβάλει 13 τροπολογίες στην πρόταση αυτή της Νομικής Επιτροπής. Μερικές είναι τεχνικού χαρακτήρα και άλλες όχι. Υπογραμμίζουν για παράδειγμα το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα δικά τους συμφέροντα, που και αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με τα θέματα που εξετάζει η δικιά μας Επιτροπή. Έπειτα υπάρχουν και δημοσιονομικές πτυχές σε αυτή την πρόταση. Γιατί οι συντάκτες του κανονισμού ισχυρίζονται ότι η μεταφορά του παρατηρητηρίου στο Αλικάντε και εφόσον αυτό τελικά ε, με το Γραφείο Ενερμόνησης, αυτό το δεύτερο έχει 400 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι μου λένε. Πλεόνασμα. Πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι το παρατηρητήριο συντηρείται από χρήματα που δίνουν και επιχειρήσεις. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει αύξηση, εφόσον υπάρχει πλεόνασμα μετά από πέντε χρόνια. Αυτή η λύση δεν θα έπρεπε να προχωρήσει και τα δημοσιονομικά ζητήματα δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν είναι κυρίως από χρήματα των επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθεί τελικά η όποια αύξηση του προπολογισμού. Θα ήταν κακή λύση αυτή. Ένα άλλο ζήτημα είναι κάτι πρακτικό που έχει να κάνει με το γεγονός ότι μεταφέρουμε το παρατηρητήριο από τις Βρυξέλλες όπου οι Βρυξέλλες συνδέονται πολύ καλά με τον υπόλοιπο κόσμο και το πάμε στο Λικάντε. Οι κάτοικοι του Αλικάντε μπορεί να το θέλουν αλλά όπως και να το κάνουμε, χωρίς να θέλουμε να τους προσβάλλουμε, είναι στην περιφέρεια. Οπότε δεν ξέρω πώς οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και πώς οι επιχειρηματίες θα μπορούν να έχουν επαφή με αυτό. Οι κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την εγγύηση ότι θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με εκπροσώπους του παρατηρητητή, όποτε το επιθυμούν με εύκολο τρόπο. Εγώ ήμουν σίγουρο ότι θα διατηρήσει ένα σημείο επαφή στις Βρυξέλλες το παρατηρητήριο. Και ελπίζω όντω να γίνει αυτό, θα είναι πολύ θετικό. Τελικά όμως, στην γνωμοδότησή μας πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτήν την ιδέα, ότι δηλαδή αυτό το σημείο επαφή της Βρυξέλλες πρέπει να διατηρηθεί για πάρα πολύ καιρό. Κάτι άλλο είναι η συνεργασία με τις δικήσεις των κρατών μελών, με τις τοπικές υπηρεσίες και τη δίκηση γενικότερα. Και αυτό το αναφέρω σε κάποια τροπολογία μου. Για να συνοψίσω λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιο γνωμοδότησή μου και από εδώ και πέρα περιμένω τις δικές σας παρατηρήσεις των σχεδόν εισηγητών κλπ. Ό,τι θέλετε για να συνεργαστούμε είμαι στη διάθεσή σας και ελπίζω να ολοκληρώσουμε το έργο μας έγκαιρα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπιέλαν για τις εξηγήσει σας. Όλοι οι σκιώδεις είναι εδώ τώρα και η κυρία Μπάστος. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι. And I also have Mr. Schwab who wanted to speak as well. Ο κύριος Schwab έχει ζητήσει το λόγο. And Mr. Repo are here. I don't know whether they want to speak also, but they're very... Εδώ είναι και άλλοι συνάδελφοι, όπως ο κύριος Repo. Did you want to um, just to start? I'm very pleased. Μπάστος. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι αλήθεια ότι δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω την ε, παρουσίαση της γνωμοδότησης από την αρχή, αλλά νομίζω ότι το κομμάτι που άκουσα με ικανοποιεί. Το προσχέδιο αυτό φαίνεται στην ουσία να περιλαμβάνει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν μια πλήρης παρουσίαση των πλέον εκτιμάτων και μειονεκτημάτων της μεταφοράς του παρατηρητηρίου στο Ινστιτούτο το οποίο λειτουργεί στο Αλικάντε. Υπάρχει ήδη λοιπόν μια αξιολόγηση του αντικτύπου η οποία δείχνει ότι η μεταφορά αυτή δεν θα υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου των προϊόντων που μας ενδιαφέρουν και θα βοηθήσει πάντα στην καταπολέμηση της πειρατείας και των, ε, και των πλαστών προϊόντων. Ταυτόχρονα λοιπόν θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε και αρκετό δημόσιο χρήμα, κάτι το οποίο δεν είναι δευτερεύον και στη συγκεκριμένη περίπτωση και γενικότερα. Δεν υπάρχουν λοιπόν πραγματικές αντιρρήσεις, δεν υπάρχουν ε, ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση με το μήνυμα το οποίο στέλνει ο εισηγητής. Μετά από συναντήσεις, τις οποίες ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πριν από το να λάβουμε την τελική ε, διατύπωση. Πριν παρουσιάσουμε λοιπόν ε, την τροπολογία, ελπίζω να μπορέσω και εγώ να βοηθήσω στη διαδικασία και να κλείσει η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε εδώ και τον κύριο Αβάνσκι από την Πολωνική Προεδρία. Ξέχασα να τον καλωσορίσω, θα του ζητήσουμε να πάρει το λόγο αργότερα αν το επιθυμεί. Κυρία Βερνιό, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Μπιέλαν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την έκθεση του κυρίου Μπιέλαν. Μπορεί να προσυπογράψω και όλες τις τροπολογίες. Κάνατε μια εξαιρετική δουλειά. Έχω και εγώ κάποια ερωτηματικά βέβαια που ταυτίζονται με τα δικά σας και τα οποία θα έλεγα έχουν σχέση περισσότερο με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αρχή αυτού του παρατηρητηρίου για την καταπολέμηση των πλαστών προϊόντων, την διάδοση των χρηστών πρακτικών, την κατάρτιση των υπευθύνων υπαλλήλων, ε, να μοιραστεί με την υπηρεσία την εξωτερική. Είναι καλό να προσπαθήσουμε με πολλούς τρόπους να προστατεύσουμε γενικά τη δημόσια υγεία γενικότερα και το συμφέρον του καταναλωτή. Θα ήθελα όμως να μας δώσουν ξεκάθαρα τη μελλοντική σύνθεση του οργανισμού αυτού. Γιατί αν πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κάνει μια ουδέτερη δημοσιονομικά αλλαγή και ταυτόχρονα να διευρύνει το πεδίο αρμοδιότητας, πώς θα γίνει αυτό, αυτή η διεύρυνση αρμοδιότητας χωρίς ε, τον να ζητηθούν επιπλέον χρήματα. Συνεπώς λοιπόν θα ήθελα να ξέρω αν αυτή η μεταφορά θα είναι κάτι το οποίο πράγματι θα ενισχύσει τις δραστηριότητές μας, αν θα καλύψει μόνο τις ανάγκες της γραμματείας, αν θα υπάρξει μια μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης μόνο προς τον ιδιωτικό τομέα, όπως κάποιες, ε, κάποια σημεία της παρουσίας της Επιτροπής αφήνουν να εννοηθεί. Αυτό μας απασχολεί. Θα ήθελα επίσης να μάθω ακριβώς τι εννοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν λέει ότι η υπηρεσία θα πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε να εκπροσωπούνται οι, πλέον θυγόμενοι οικονομικοί τομείς από τις επιθέσεις στα πνευματικά δικαιώματα βλέποντας το πόσο λίγα έγγραφα έχουμε στη διάθεσή μας, πώς μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι φύγονται περισσότερο. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός τομέων που φύγονται. Και αυτό το οποίο φοβάμαι είναι να μας πούνε μετά ότι θα πρέπει να συμμετέχουν αυτοί οι οποίοι κατέχουν τα δικαιώματα και αυτοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες και μέσω του διαδικτύου. Λέει επίσης το κείμενο ότι θα πρέπει να υπάρξει εκπροσώπηση και των, θα πρέπει να υπάρξει εκπροσώπηση των μικρομεσαίων και των καταναλωτών. Νομίζω, εν πάση περιπτώσει, λέει η κυρία Δερνιό, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στους οικονομικούς τομείς οι οποίοι θίγονται από την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, από τους παροχείς στο διαδίκτυο και από την παρουσία των καταναλωτών και των μικρομεσαίων. Ένα κομμάτι δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κειμένου της πρέπει να γίνει αντικείμενο ενίσχυσης. Πάντα για το κείμενο της Επιτροπής ένα άλλο αρνητικό είναι ότι δεν θα πρέπει να βάλουμε στο ίδιο επίπεδο το θέμα της πειρατείας από τη μία και το θέμα των πλαστών προϊόντων από την άλλη. Μιλάμε πολύ για πειρατεία, αλλά νομίζω ότι τα πλαστά προϊόντα δημιουργούν πολύ περισσότερα προβλήματα και δεν εμπλέκονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές δεν, ξε, δεν διευκρινίζεται αυτό στο κείμενο και δεν δίδονται οι ίδιες απαντήσεις στα δύο διαφορετικά φαινόμενα. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ζητήσω να υπάρξει διάλογος και με την Γενική Διεύθυνση ΚΟΜ και όχι μόνο με την Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΚ για την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την εξοικονόμηση και την ασφάλεια. Αν πράγματι θέλουμε να προχωρήσει η εσωτερική αγορά, δεν μπορούμε να αρνηθούμε και δεν το αρνούμε εγώ τις συνέπειες της πειρατείας πολιτιστικών αγαθών. Αλλά δεν θα πρέπει να προωθήσουμε ένα κείμενο μόνο προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν και άλλες πλευρές ενδιαφέρουσες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για τους μικρομεσαίους και τους πολίτες και καταναλωτές και η έκθεση φαίνεται να υποτιμά αυτό το κομμάτι. Αυτό πρέπει να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των συζητήσεων που έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό και που κάναμε και στο φόρουμ της Κακοβίας άλλωστε. Και να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον κύριο Μπιέλαν. Είναι σαφές ότι έχετε τα ίδια ερωτηματικά με μένα. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Πράγματι, Βλέπω ότι οι μικρομεσαίες και οι καταναλωτές προβλέπεται να είναι στις αντιπροσωπευτικές συναντήσεις του παρατηρητηρίου. Υπάρχουν όμως και θέματα παρουσίας των κυβερνήσεων. Ο κύριος Μπίλαν έχει κάνει πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή και μένει ακόμα όμως να διευκρινίσουμε αρκετά. Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε να ευχαριστήσω τον κύριο Πίελαν για την έκθεσή του. Δεν είναι πολύ αμφιλεγόμενα τα πράγματα, οπότε θα είμαι σύντομος. Ξέρουμε όλοι το πρόβλημα της πειρατείας, της παραποίησης, που βλάπτει άμεσα την οικονομία, αλλά και τον καταναλωτή και βεβαίως δημιουργεί προσκόμματα για την κοινοτομία. Η δημιουργία του παρατηρητηρίου ήταν ένα πολύ καλό βήμα. Τώρα πρέπει να προχωρήσει και να ενισχυθεί η εργασία του. Το, το να μην χρειάζεται βεβαίω επιπλέον προπολογισμό για να γίνει αυτό είναι σαφέ ότι πρέπει να αποτελέσει μια ε, επιλογή. Η μεταφορά στο Αλικάντε νομίζω ότι δημιουργεί, μας δίνει τη δυνατότητα να μην δημιουργήσουμε μια νέα, μια νέα δομή, αλλά να συνεχίσουμε την ε, εργασία που έχει ξεκινήσει ήδη. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό ήταν σκόπιμο και σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν ο συνάδελφος Μπίλα νομίζω ότι έχει κάνει μια γνωμοδότηση πολύ ισορροπή, συμπεριλαμβάνει τους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μιλά για την λήψη των μέτρων που θα πρέπει να λάβουν τα κράτη-μέλη μιλά και για το γραφείο, της, ε, το γραφείο εναρμόνισης, το οποίο θα πρέπει να έχει την επαρκή ε, χρηματοδότηση. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά στοιχεία και τον ευχαριστώ και πάλι για την γνωμοδότησή του. Ευχαριστώ. Ε, Mr. Ο κύριος Έγκστρομ. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η κυρία Βερνιού. και την πειρατεία και την παραποίηση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο είναι το, ε, ε, το εμπορικό, η εμπορική παραποίηση και άλλο είναι το downloading, η πειρατεία. Στα πλαίσια της έκθεσης ε, η Κομισιόν ορίζει την πειρατεία ως εμπορική εισαγωγή CD και DVD που βεβαίως όλοι συμφωνούμε είναι παράνομο, θα πρέπει τέλο πάντων να είναι παράνομο και είναι επιζήμιο. Σήμερα βλέπουμε στην πρόταση της Κομισιόν να λέει ότι ε, δεν είναι εμπορική, το, η πειρατεία δεν σημαίνει εμπορική, παρα, ε, εμπορικό κατέβασμα ή εισαγωγή αυτών των CD και DVD. Θα, νομίζω ότι θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε τα δύο αυτά. Δεύτερο σχόλιο για το κονδύλιο, για τα χρήματα. Ο κύριος Μπιέλαν είπε ότι μέχρι τώρα από, το, από την ώρα που έγινε το παρατηρητήριο όντως ήταν ε, μεγάλη, ε, μεγάλη επιτυχία, ασχολήθηκε με το θέμα της, ε, των εμπορικών σημάτων. Μίλησε και για, την, για τον επιπλέον προπολογισμό που έχει παραμείνει ως πλεόνασμα στο παρατηρητήριο. Δεν άκουσα βέβαια τον ακριβή αριθμό. Αλλά ο κύριος Μπιελέν έχει δίκιο ότι τα χρήματα αυτά ε, δικαίω ανήκουν στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ε, καταχωρήσει τα εμπορικά του σήματα. Παρόλο που βρίσκονται σε κάποιο άλλο διαφορετικό ε, λογαριασμό, δεν σημαίνει ότι είναι ξαφνικά κάποια λεφτά που βρέθηκαν έτσι από το πουθενά. Και ένα τελευταίο σημείο. Δεν είναι μυστικό ότι αυτό το παρατηρητήριο θεωρώ ότι είναι πραγματικά χαμένος χρόνος και χαμένα χρήματα. Θα ήταν χρήσιμο εάν μπορούσε να συλλέγει επιστημονικά δεδομένα, αλλά δυστυχώς δεν ε, θεωρώ ότι το κάνει αυτό. Για παράδειγμα, στη δεύτερη παράγραφο του επεξηγηματικού σημειώματος, λέει ότι η έκθεση τέρα που έγινε το 2010 ε, ξεκίνησε λόγω της, ε, του αιτήματο να γίνει από ε, εμπορικά συμφέροντα. έτυχε μεγάλες κριτικής από όλους όσους την είδαν και είναι η μόνη μελέτη που αναφέρει η Κομισιόν. Δεν αναφέρει τίποτε άλλο. Έχουν γίνει πάρα πολλές ακαδημαϊκές μελέτες που είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες και έχουν πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα και στοιχεία. Και αυτό εμένα με ανησυχεί, πάντα με ανησυχούσε. Οπότε, εξεκολουθώ να πιστεύω ότι το παρατηρητήριο αυτό είναι χαμένα λεφτά και χαμένος χρόνος, οπότε δεν έχω ιδιαίτερα σχόλια να κάνω για το πώς θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του. Ευχαριστώ. Ωραία. Επομένως, Ελπίζω ότι θα υποβάλλετε τροπολογίε για την έκθεση του κύριου Μπιέλλον, αν θέλετε να βελτιωθεί σε κάποιο σημείο. Ο κύριο Σβάμπ ήθελε το λόγο και η κυρία Γκάλο ήθελε το λόγο μετά. Ο κύριο Ροπό. Όχι, ναι. Ο κύριο Σβάμπ. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχουμε τον κύριο Μπερζεβά εδώ πάλι από την Κομισιόν με νέα καθήκοντα είναι, ε, έχει εργαστεί για το παρατηρητήριο εδώ στις ε, Βρυξέλλες. Θα συμφωνήσω με τους ε, προλαλήσαντες. Έχουμε την ευκαιρία τώρα αυτό το παρατηρητήριο να το εξοπλίσουμε με, τα, με την εμπειρογνωμοσύνη και τα κονδύλια που είναι απαραίτητα για να μπορεί να κάνει επαρκώς τη δουλειά του. Το είπε και, ο συνάδελφος Έγκστρομ. Ε, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η σχέση με τις υπόλοιπε πρωτοβουλίες που υπάρχουν για την προστασία της πνευματική ιδιοκτησία Και αυτό το έχουμε πει και για την εφαρμογή του, τον, ε, για την δελωνία για την εφαρμογή του IPR. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα ακόμα εκκρεμή τα οποία πρέπει να λύσουμε. Και ελπίζω ότι το παρατηρητήριο, ειδικά μέσω της σύνδεσης με την εργασία του Γραφείου Εναρμόνισης για την Ιστορική Αγορά, θα μπορέσει να λειτουργήσει, αλλά και σε πιο στενή συνεργασία με την Κομισιόν θα μπορέσει να συμβάλλει ώστε να πέσει περισσότερο φως σε όλη αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι είναι καλό που ε, τα κορδίλια του Γραφείου Εναρμόνισης ε, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα επαναεπενδύσουμε στην αγορά. Ο συνάδελφος Μπίλεν εδώ λέει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φυσικά είμαι ανοιχτό σε αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να πούμε ότι από, από τα δικαιώματα IPR σε σχέση με το θέμα αυτό υπάρχουν πολλά προβλήματα, κυρίως για τις μεγάλες επιχειρήσεις και μάλλον αυτό θα είναι και το σημείο για το οποίο ο κύριος Έγκστρομ βλέπει έτσι πολύ σκεπτικά και με αμφιβολία στα πράγματα. Νομίζω όμως ότι το διαχωρισμό της εμπορικής χρήσης ή της ιδιωτικής χρήσης που κάναμε χτες είναι ένα σημαντικό σημείο το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Ελπίζω η Κομισιόν, και γι' αυτό κύριε Πρόεδρε είναι σημαντικό για την Επιτροπή μας, να το προχωρήσουμε, να το παρακολουθούμε, να μην θεωρήσει ότι το θέμα αυτό έχει ε, κλείσει επειδή υπάρχουν κάποια επιπλέον κονδύλια τα οποία βρίσκονται εκτός του προπολογισμού που έχει προβλέψει η Κομισιόν. Νομίζω ότι αυτό, το, αυτή την έκθεση θα πρέπει να την δει πάρα πολύ προσεκτικά, θα πρέπει να ασχοληθεί με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και να δώσει τα απαραίτητα κονδύλια έτσι ώστε να μπορέσουν να προκύψουν και καλές προτάσεις. Γιατί νομίζω ότι στην Ευρώπη θα, είμαστε, ε, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την καινοτομία μας και οικονομικά στο μέλλον, μόνο αν υπάρχουν ιδέε που μπορούν να προωθηθούν εύκολα. Μόνο έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε την πραγματική ιδιοκτησία. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε αυτή την ε, έκθεση, ώστε, να την, ώστε αυτή την έκθεση να την προωθήσουμε ε, με, και να την εμπλουτίσουμε με τέτοια στοιχεία ώστε να μπορέσει να γίνει αποδεκτή στο τέλο. Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η πρόταση γιατί είναι πραγματικά α, πάρα πολύ σημαντική ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Γκάλου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι έχοντας ακούσει τον συνάδελφο Άγκστρομ, έχω την εντύπωση ότι κάπου το έχουμε όχι ξαναδεί, αλλά ξανακούσει. 18 μήνες πίσω δηλαδή ένιωσα ότι πήγα, γιατί είναι αυτές οι ατέρμονες συζητήσεις που κάνουμε και που λέμε ότι τα πλαστά δεν είναι το ίδιο με την πειρατεία και ότι πρέπει να τα εξετάζουμε διαφορετικά. Σήμερα στην νομική επιτροπή που είναι και η αρμόδια επί της ουσίας και με τον συνάδελφο Ιτάλγο που είναι σοσιαλιστής καταλήξαμε σε συμφωνία για αυτά τα θέματα διότι τα βάζουμε με το παρατηρητήριο και λέμε ότι δεν έκανε τίποτα και ότι δεν μπόρεσε να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία. Μα ακριβώς είναι γι' αυτό ότι τον συγχωνεύουμε τώρα και έτσι θα έχουμε τα μέσα να έχουμε πραγματικές μελέτες. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν συγχρόνως να λέμε ότι χρειαζόμαστε νούμερα για να κρίνουμε τη ζημιά που γίνεται τόσο από τα πλαστά όσο και από την πειρατεία που θέλουμε να τα διακρίνουμε, εντάξει, το καταλαβαίνω, και συγχρόνως να λέμε ναι, ότι δεν βελτιώνουμε τα μέσα προκειμένου να το πετύχουμε αυτό. Αυτές είναι οι δικές μου οι παρατηρήσεις. Εγώ πιστεύω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει και πιστεύω ότι δεν πρέπει να συνεχίζουμε ισαΐ αυτό το σημειωτόν που κάνουμε χωρίς να προχωράμε. Ας προχωρήσουμε. Είναι προς το συμφέρον όλων μας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν πρέπει να παρετούμαστε, να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και να μην κάνουμε τίποτα. Πράγματι. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή, ιδίως όταν πρόκειται για την προστασία του καταναλωτή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα προϊόντα στην αγορά και μερικές φορές δεν είναι ασφαλή. Να φροντίσουμε να έχουμε λοιπόν αρκετού πόρου και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε κονδύλια. Λοιπόν, συμφωνώ με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμεί. Άλλο κανεί. Ένα σχόλιο έχω εγώ από τη δικιά μας την πλευρά. Για την γενική εποπτεία και τη στρατηγική του παρατηρητήριου. Εδώ βλέπω ότι οι συναντήσεις θα είναι ανοιχτές στο παρατηρητήριο. Καλό αυτό. Αλλά προβλέπετε κάποιο ε, συμβούλιο, κάποιοι εμπειρογνώμονες που να συμβουλεύουν για τα προγράμματα έρευνας και για το τι μελέτες πρέπει να αναλαμβάνει το παρατηρητήριο. Πώς ε, θα γίνεται ή θα είναι το γραφείο αναρμόνησης που θα το λέει. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό για μένα. Έπειτα εγώ καταλαβαίνω βέβαια αυτό που λέει ο Κρίστεν Άμστρομ όσον αφορά τον ορισμό της πειρατεία. Καταλαβαίνω τι λέει και τι εννοεί. Είναι μεν στον τίτλο, αλλά όχι τόσο στο περιεχόμενο της πρότασης. Νομίζω λοιπόν ότι το πρώτο που είναι σημαντικό είναι η διαφάνεια αλλά και για τις ομάδες ενδιαφερομένων, καλό θα ήταν να μπορούν και αυτοί να προτείνουν ιδέες για έρευνες, για μελέτες. Και η κυρία Μπανιούλ είπε πολύ σωστά ότι πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί των οποίων τα συμφέροντα επηρέαζονται περισσότερα, γιατί ίσως οι έρευνες να δείξουν ότι ορισμένοι, ορισμένο τα συμφέροντα δεν λαμβάνονται υπόψη καθόλου, οι άλλων περισσότερο και άλλο λιγότερο. Οπότε, να και το άλλο θέμα είναι οι αγορές online και εκεί τα πλαστά, είτε πρόκειται για ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αεροσκαφών, άλλα αγαθά και τους καταναλωτές, τρόφιμα, φάρμακα και και και Ελπίζω το παρατηρητήριο λοιπόν αυτό να ασχοληθεί με το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας ευρύτερα και όχι περιοριστικά. Και όχι μόνο για το τι κατεβάζει κανείς μέσω του διαδικτύου. Λοιπόν, ο κύριος Μπέντσεμον, ο κύριος Βάνσκι, για το πώς έχουμε προχωρήσει το Συμβούλιο και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπίλαν βεβαίως πάντα για να μας πει ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα και να κλείσουμε έτσι τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, εξετάζουμε με ικανοποίηση την έκθεση του κυρίου Μπίλαν όπως επίσης και το γεγονός ότι έχει γνωμοδοτήσει, θα γνωμοδοτήσει η δικιά σας η Επιτροπή που ασχολείται με την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών. Οπότε θα έχουμε και αυτή την οπτική γωνία. Κάποια γενικά σχόλια θα κάνω προσπαθώντας να απαντήσω στις παρατηρήσεις σας. Πρώτον, το πιο εύκολο ίσως είναι η ανησυχία σας αυτή για το, ότι το Αλικάντε είναι μακριά από τις Βρυξέλλες και όταν θα γίνονται συνεδριάσεις στο παρατηρητήριο δεν θα μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση ενδιαφερόμενοι. Η υπηρεσία εκεί έχει δεσμευτεί να οργανώνει και στις Βεξέλλες συνεδριάσεις, ακριβώς για αυτό το σκοπό. Οπότε νομίζω ότι αφού υπάρχει αυτή η δέσμευση θα τηρηθεί, δεν θα την είχαν κάνει αν δεν ήταν κάτι το εφικτό. Έπειτα έρχομαι στο θέμα της εκπροσώπησης των διαφόρων ομάδων στο παρατηρητήριο. Μέχρι τώρα το παρατηρητήριο είχε τη δικιά του δυναμική. Υπάρχει εκπροσώπηση των καταναλωτών και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί. Για να είμαστε ειλικρινεί, συμφωνούμε με την άποψή σα και εμεί πιστεύουμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι με του οποίου συζητάμε πρέπει να συμμετέχουν κατάσταση είναι ότι έχουμε καλέσει ομοσπονδίες μέχρι τώρα και όχι ατομικά επιχειρήσεις. Με το σκεπτικό ότι οι ομοσπονδίες εκπροσωπούν όλες τις επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες. Αλλά σημειώνω αυτό που λέτε ότι για τις μικρομεσαίες έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή τους. Δεν θέλουμε όμως να το επισημοποιήσουμε γιατί μπορούμε να φανταστούμε ότι για διαφορετικά θέματα θα χρειάζεται διαφορετική εκπροσώπηση. Αλλά κατά τη μεταβατική περίοδο, αν με τι άλλο, θα κοιτάξουμε τη σύνθεση και νομίζω ότι η διαφάνεια που ζητάτε θα δείτε ότι υπάρχει στην πρότασή μας. Θα αναπτυχθεί περισσότερο και κάθε χρόνο θα υπάρχει κάποιο πρόγραμμα εργασίας μπορεί να καταλήξει σε αιτήσια έκθεση ώστε να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια όπως ζητήσατε εδώ. Για τον προπολογισμό. Τι θα γίνει με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις, πώς θα ρυθμίζονται. Αυτό θα διευκρινιστεί στο πρόγραμμα εργασίας. Θα έλεγα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ ότι δεν υπάρχει πρόθεση αύξησης των ε, απαιτήσεων του Γραφείου Αναρμόνησης, αλλά αυτό που πιστεύουμε εμείς είναι ότι πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες. Και όλα αυτά που λέτε ότι πρόκειται για χρήματα των μικρομεσαίων για να καταχωρήσουν εμπορικά σήματα, Από τους έξι μήνες που έχω παρακολουθήσει το παρατηρητήριο μπορώ να σας πω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούν ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται και το παρακολουθούν. Τώρα για τη χρήση της λέξης πειρατεία. Όσο το παρατήριο προχωράει υπάρχει μια ισορροπία με το θέμα των παραπημένων προϊόντων. Υπάρχουν πολλές ομοσπονδίες και συμμετέχουν. Πάντως έχετε δίκιο πρόεδρε για αυτό που λέτε, ότι πιο πολύ ασχολούμαστε με το πώς να κατεβάσουμε μέσω του διαδικτύου ε, προϊόντα. Πάντως το θέμα της πειρατείας είναι σημαντικό να έχει συγκεκριμένο και σωστό ορισμό. Το παρατήριο έχει ασχοληθεί πάντως γενικά με τις παραβιάσεις και τη συμμόρφωση. Ο σκοπός του δεν είναι να επικεντρωθεί περισσότερο στον ένα ή στον άλλο τομέα. Τέλος, για τις προτεραιότητες. Βλέπετε δύο πράγματα στην έκθεση. Πρώτον, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμείς θα θέλαμε να μπορούμε να ζητήσουμε και να έχουμε συστάσεις από το ίδιο το παρατηρητήριο. Έτσι ώστε να υπάρχει κατεύθυνση και από εμά και από το Κοινοβούλιο. Βλέπετε ότι θα μπορούσαν κάποιοι από το Κοινοβούλιο να ασχολούνται με το παρατηρητήριο, να εμπλέκονται, ώστε να υπάρχει και μια πολιτική διάσταση μέσα αλλά και για τη δυναμική. Προς το παρόν, το παρατηρητήριο ε, ακολουθεί πολύ τους εμπειρογνώμονες και τους εκπροσώπους των κρατών ε, μελών, τα αντίστοιχα γραφεία δηλαδή σε εθνικό επίπεδο. Η σημερινή σύνθεση είναι τέτοια που το παρατηρητήριο συνεδριάζει με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση. Και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών συνεδριάζουν χωριστά, μερικές φορές βέβαια και όλοι μαζί. Οι συναντήσεις αυτές των κρατών μελών είναι κάτι που έχει συμφωνηθεί από το πρόγραμμα εργασίας. Μέχρι τώρα πάντως έχει προχωρήσει καλά αυτή η μορφή. Βέβαια με τον νέο κανονισμό θα βελτιωθεί η διαφάνεια και θα έχουμε καλύτερους πόρους. Το θέμα αυτό πάντως της διακυβέρνησης μέχρι τώρα έχει λειτουργήσει καλά και θέλουμε να συνεχίσει έτσι. Το θέμα δεν είναι ποιο θα γείται, αν θα είναι η Επιτροπή ή όχι. Είναι οι εμπειρογνώμονε μέσα από το παρατηρητήριο που ηγούνται. Και κάτι ακόμα. Χάρη στο παρατηρητήριο έχουμε αναλάβει μια μεγάλη μελέτη με την εταιρεία Grant και θέλω να σας διαβεβαιώσω και ευχαρίστω να το συστήσω μαζί σας και μετά έχουν αναθεωρήσει, αναθεωρήσει όλες τις μελέτες, 200 και συνεχίζουν να δουλεύουν πάνω σε αυτές. Γιατί? Για να δούνε ποια θα είναι τελικά μια αξιόπιστη μεθοδολογία προκειμένου να μπορούμε να έχουμε αριθμητικά αποτελέσματα για την πειρατεία και, και την παραποίηση. Η μελέτη αυτή θα είναι έτοιμη στα τέλη της χρονιάς. Έγκαιρα δηλαδή. Είναι προτεραιότητα για το παρατηρητήριο, πρέπει να ξέρετε τα μέλη του παρατηρητηρίου. Έτσι λένε ότι είναι προτεραιότητα για αυτούς γιατί χρειάζεται ακόμα και οι ενδιαφερόμενοι, η βιομηχανία, οι διάφοροι κλάδοι το θέλουν. Θέλουν να έχουν, όπως είπε και η κυρία Λεκό, χρειάζονται συγκεκριμένα στοιχεία, αν μη τι άλλο εκτιμήσεις πάνω στις οποίες να συμφωνούν όλοι. Οπότε οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι τροπολογίες που βρίσκω πολύ καλές γιατί έτσι το παρατηρητήριο θα μπορέσει να βοηθήσει τους πολιτικούς να υιοθετήσουν ε, την μελλοντική πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που δώσατε κάποιες απαντήσεις και για την προσφορά σας να ενημερώσετε ακόμα περισσότερο τα μέλη. Κυρία Μπάνσκι της Πολωνικής Προεδρίας, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για την πρόοδο στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπιάλαν, τον εισηγητή, για μια εξαιρετική έκθεση που ε, ενημερώνει αρκετά σε κάποιους τομείς. Να σας ενημερώσω και εγώ με τη σειρά μου ότι έχει υπάρξει πρόοδο στο Συμβούλιο. Υπάρχει πλέον συνένεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη σχετικά με την αρχή Αποδοχή των συμβιβαστικών προτάσεων της Προεδρίας. Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν στην ομάδα εργασίας την Αυμόδια τον μήνα Σεπτέμβριο. Δεν πρόκειται για την τελική πρόταση βέβαια του Συμβουλίου ακόμη. Νομίζω όμως ότι σε 15 περίπου μέρες θα μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε την επόμενη πρόταση της Προεδρίας. Οι αλλαγές τις οποίες θα προτείνουμε θα έχουν σαν στόχο στην καλύτερη εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων του συγκεκριμένου οργάνου, έτσι ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Θέλουμε να υπάρχει επίσης και ευελιξία σχετικά με τα κατεπήγοντα θέματα, Ανάμεσα στα δύο όργανα πρέπει να βελτιωθεί η επικοινωνία και η ουσιαστική διαχείριση της υπηρεσίας αυτής, ιδιαίτερα γύρω από τις λεγόμενες νέες αποστολές. Πάντως έχει υπάρξει, επαναλαμβάνω, πρόεδρος στο Συμβούλιο και ελπίζω ότι ήδη από εφέτος θα ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα επιπλέον μικρό σχόλιο για την έδρα του παρατηρητηρίου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, θα πρέπει να παραμείνει σε μία και να συνεδριάζει σε μία έδρα το συγκεκριμένο παρατηρητήριο. Αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Το παρατηρητήριο δεν είναι στατικό και μετακινείται κατά κάποιο τρόπο. Συνεδριάζει σε πολλά μέρη μεταξύ των οποίων και Βρυξέλλες. Πραγματι η συνεισφορά του Συμβουλίου φαίνεται από την τελευταία σας παρατήρηση, λέει ο Πρόεδρος. Κύριο Μπιέλαν, μπορείτε να κλείσετε τη συζήτηση και να μας επιβεβαιώσετε το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια των συναδέλφων της Επιτροπής. Νομίζω ότι τα σχόλια ήταν υποβοηθητικά και επικοδομητικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βερνιό. Έθεσε πάρα πολλές ερωτήσεις, οι οποίες απευθύνονταν κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να ικανοποιήθηκε η κυρία Βερνιό από τις απαντήσεις της Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά συμμερίζομαι τις ανησυχίες της κυρίας Βερνιό σε πάρα πολλά θέματα. Υπόσχομαι ότι θα έλθω σε επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές και από εδώ και πέρα και με όλα τα μέλη της Επιτροπής άλλωστε που ενδιαφέρονται για αυτή τη γνωμοδότηση. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα. Από ό,τι γνωρίζω τα πράγματα έχουν ως εξής. Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 12η μεσημβρινή μπορείτε να καταθέσετε τις τροπολογίες σας. Έχετε δύο εβδομάδες. Θα εξεταστούν οι ε, τροπολογίες αυτές στη συνεδρία μας της 22ης Νοεμβρίου και ταυτόχρονα θα υπάρξει και ψηφοφορία. Η γνωμοδότηση θα πρέπει να γίνει δεκτή από την Επιτροπή Γιούρη στη συνέχεια μέσα στο Δεκέμβριο. Φέτος δηλαδή όλα αυτά έτσι ώστε η ψηφοφορία να μπορέσει να γίνει στις 16 Ιανουαρίου του 2012 στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ όλους για την βοήθειά σας και ελπίζω ότι θα συνεχίσω ε, την επικοινωνία μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέλλαν. Ήταν εξαιρετική συζήτηση θα υπάρξει μια μικρή διακοπή μέχρι τις 10, οπότε θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες για τις τρεις προτάσεις που έχουμε, Κρόιτσμαν, Λεγκρίπ και Ράπτη. Θα χρειαστείτε τις ε, κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Διακόπτουμε λοιπόν μέχρι τις 10.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

Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όσους δεν χαιρέτησα πιο πριν. Έγιναν πολύ ωραίες ε, συζητήσεις το πρωί για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο. Πάμε στις ψηφοφορίες μας. Έχουμε τρεις ψηφοφορίες για σήμερα. θα φροντίσω να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην χάσουμε οποιαδήποτε τροπολογία ή συμβαστική τροπολογία. Να δώσω το λόγο πρώτο στον κύριο Κρόιτσμαν. Πριν ξεκινήσουμε την έκθεσή του για τον online τζόγο, να μας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές για την ε, πολύ καλή συνεργασία μας. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, καταλήξαμε σε πολλές συμβιβαστικέ τροπολογίες και νομίζω ότι πλέον έχουμε μία γνωμοδότηση για τον ε, τζόγο online που θα μπορέσει να τύχει ε, της συμφωνίας και του Κοινοβουλίου. Όταν θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια η πρώτη θέση μου ήταν να έχουμε μεγάλη πλειοψηφία, ευρεία πλειοψηφία γιατί όλοι είναι πεπισμένοι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Υπάρχει αρκετό κατακαιρματισμό. Προσπαθούμε να λύσουμε λοιπόν όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Ευχαριστώ για πάλι όλου του ε, σκιώδει που συνεργάστηκαν μαζί μου. Δουλέψατε όντω πολύ σκληρά για να καταλήξετε σε αυτή την πρόταση και σα ευχαριστούμε κύριε Κρόιτσμαν. Πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Πάμε στην νέα παράγραφο 1α. Τροπολογία 71. Υπέρ. Μπορεί να πρέπει να το δούμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία για την ε, τροπολογία 71. Παράγραφος 1α, καινούρια. Uh, Έχετε βάλει όλοι τις κάρτες σας για να ψηφίσετε. Right. Ωραία. 33 κάρτες υπάρχουν, 32 έχουν ψηφίσει. Κάποιος δεν έχει ψηφίσει. 33 έχουν τοποθετήσει τις κάρτες τους, κάποιος δεν έχει ψηφίσει όμως. Μήπως δεν δουλεύει κάποιο, κάποια συσκευή, όχι, εντάξει. Uh, no, I'm not, όχι, όχι, εγώ δεν ψηφίζω. Υπάρχουν τρία, τρία μέλη τη ομάδα μου. Εν πάση δεν ξέρω ποιο ε, δεν έχει ψηφίσει. Α, ωραία. Εντάξει. 32 λοιπόν υπέρ και μία ψήφο κατά. Οπότε εγκρίνεται η τροπολογία. Οπότε, τώρα, οι υπόλοιπε κατά Πιπτούν Πάμε στην Γιούρι 11, στο αντίστοιχο σημείο. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Σε 72. Ρόσφορ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία 70 του Hans Πέτερ Μάιερ ως ε, προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στην έκον. Όλα αυτά πάλι είναι με τμήματα που συνδέονται. Έκον 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έκον. Αντίστοιχο τμήμα 2. Υπέρ. Α, συγγνώμη, καλύπτεται από την παράγραφο 1. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Πάμε στην 13. Κύριο Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της ε, τροπολογίας του κυρίου Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται. Πάμε στην 73. Δεν την ψηφίζουμε όμως, νομίζω. Πάμε στην 75 του κυρίου Γιόνγκ, Υπέρ. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε ηλεκτρονικά. Άρχιδε η ψηφοφορία για την τροπολογία 75. Uh, the vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11 προς 23. Πάμε στην 78 του κυρίου Χουάν Νόγκ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 81 από αρκετούς συναδέλφους. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 79 ως προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 79. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 προς 21. 80. Πάλι Χουαγνόγκ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 85 Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οι 83 και οι 84 καλύπτονται. 82 του κυρίου Χουαγνόγκ. Ως προσθήκη και πάλι. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 82. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15 προς 20. 86. Πάλι, πάλι Νόγκ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 86. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 προς 20. 20. Η 87 νομίζω καταπίπτει. Σωστά. Όχι. Όχι, θα την ψηφίσουμε την 87. 87 λοιπόν του κυρίου Ταραμπέλα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 88. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι. Ποιο είναι υπέρ για την 88. Κατά. Απορρίπτεται. 89. Άρχεται η ψηφοφορία για την 89. The vote's closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15 προς 20. Τροπολογία 90. Αμπάντ και λυπή. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 91, η 91 καταπίπτει. Πάμε στην 92. Άρχεται η ψηφοφορία για την 92. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 18 προς 15. 95. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 94 της κυρίας Σεναλόβα. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 93 δεν την ψηφίζουμε, είναι γλωσσική τροποποίηση. Πάμε στην 96. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 97. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 97. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24 προς 10. Τροπολογία 199 μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 98 ως προσθήκη. Υπέρ. Νομίζω ότι θα την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 98. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 προς 11. 101 ως προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία για την 101. Πέρας. Απορρίπτεται. 4 προς 31. 102. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην ε, τροπολογία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 108. Υπέρ υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Γιούρι 7, υπέρ, κατά, αποχές, δεν κοίταγα, συγγνώμη, να την δούμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την Γιούρι 7. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 5 προς 16. 109 για τις κυρίες Αναλόβα. Άρχεται η ψηφοφορία για την 109. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11 προς 23. Πάμε στην 113, κύριο Κέλλη. Άρχεται η ψηφοφορία για την 113. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 προς 14. Η 110 καταπίπτει, άρα... Α, όχι. Η 110 πρέπει να την ψηφίσουμε. 110 λοιπόν. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 110. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 προς 10. Έπρεπε να την ψηφίσουμε τελικά την 110. 114 και 115 και αυτές πρέπει να τις ψηφίσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, 114 και 115. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 112 του κυρίου Κάρας. Άρχεται η ψηφοφορία για την 112. Πέρας. Εγκρίνεται. 25 προς 11. 111 καταπίπτει. Έκον 6. Υπέρ. Να το δούμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την ε, τροπολογία Έκον 6 πέρα. Εγκρίνεται. 20 προς 14. 117. Μάντερς. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Χαίρομαι που είστε εδώ κύριε Μάντερς. Πάνω στην ώρα ήρθατε που απορρέφθηκε η τροπολογία σας. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 127 του κυρίου Γκρέκ. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 138 του κυρίου Χουαγνόκ. Υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. Εκον 3. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για την Εκον 3. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16 προς 18. Πάμε στη Γιούρι 3. Γιουριένα. Γιουριένα, Γιουριένα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Θα το δούμε και τις υπόλοιπες. Λοιπόν, 140 και 141. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Γιούρι 4. Καλύπτεται. Η... Ναι, καλύπτεται. Αλλά πρέπει να την ψηφίσουμε. Α, είναι η ίδια. Μάλιστα. Πάμε στην 116 του κυρίου Φιέλνερ. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 116. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 προς 10. Πάμε στην 23 η οποία καταπίπτει. 139 του κυρίου Πουπάκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην, τροπο, στην συμβαστική τροπολογία 11 για την παράγραφο 9. Συμβαστική τροπολογία 11. Συμβαστική 11 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε την 176 που είναι αρκετές, αρκετές λίγες πιο πίσω από τον κύριο Γκρέκ παράγραφος 9α καινούρια άρχεται η ψηφοφορία για την 176 πέρας εγκρίνεται 176 εγκρίνεται 25 προς 10 συμβαστική 10 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 187. Του κυρίου Ντεγιόγκ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 186. Μπουσούτλ και Ελυπή. Ως προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία για την 186. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 προς 10. 192. Σάλντε Μόζα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 190 και 191 δεν τις ψηφίζουμε. Γιούρι 10. Γιούρι 10. Άρχεται ψηφοφορία για τη Γιούρι 10. Πέρας. Μπορείτε να επιταχύνετε λίγο. Εγκρίνεται. 18 προς 15. 193 την ψηφίζουμε. 193 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία για την 193. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 προς 10. Γιούρι 12. Υπέρ. Αν θα την ψηφίσουμε και αυτή ηλεκτρονικά. Γιώρι 12. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 προς 15. Πάμε στην παράγραφο 12. Υπάρχουν ταυτόσιμες ε, τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία για την 195, 196 και 197. Πέρας. Απορρίπτονται όλες. 10 προ 21. 198 του κυρίου Γκρέχ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 2.25 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Την εικόν 7 την έχει καλύψει ήδη η 2.25. Εκόν 8. Νέα α, παράγραφος 13α. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έκον 9. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Εκόν 13. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 223. Υπέρ κατά, εγκρίνεται. Έκον 15 ως προσθήκη. Ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην Γιούρι 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14. 2.16 του κυρίου Κέλλη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2.17. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2.18. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 2.18. Πέρας. Το ΕΛΚ έχει έναν επιπλέον. Κάποιος ήρθε από το ΕΛΚ. Μια, μπορεί να βγει μια κάρτα παρακαλώ. Ωραία, εντάξει. Πέρασε. Εγκρίνεται. 25 προς 10. 2.15. Σολτεμόζα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2.14. Της κυρίας για Τενμάκη και άλλων. 2.14. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 2.14. Πέρας. Εγκρίνεται. 18 προς 17. Έκον, το δεύτερο κομμάτι της έκον 11 ε, δεν το ψηφίζουμε. Πάμε στην έκον 11, αντίστοιχο τμήμα 1. Υπέρ. Υπέρ της έκον 11. Κατά εγκρίνεται. 2.19. Άρχεται η ψηφοφορία για το 2.19. Πέρας. Απορρίπτεται. 14 προς 21. 2.24. Άρχεται η ψηφοφορία για το 2.24. Πέρας. Απορρίπτεται. 13 προς 21. 2.20. Υπέρ. Ε, άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρας. Απορρίπτεται επίσης. 2.22. Άρχεται ψηφοφορία για το 222. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.27. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2.28. Η 2.28 καταπίπτει. Πάμε στη συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται. Πάμε στην 2.37. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 2.37. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.42 της κυρίας Κόμη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 2.41 του κύριου Πιτέλα, υπέρ, κατά, επίσης εγκρίνεται. Συμβαστική 16, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάμε στην 2.45 του κυρίου Φιέλνερ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 2.45. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται. Πάμε στην 226 του κυρίου Κάρας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 261 του κυρίου Χουάνγκ Η, η ψηφοφορία για τη 261. Πέρας. Εγκρίνεται. 262 της κυρίας Χέντ. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 262. Πέρας. Απορρίπτεται. 260 της κυρίας Χέντ. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 260. Πέρας. Απορρίπτεται. Έκον 19. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 272 Φιέλνερ. 272 Φιέλνερ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 13 του κυρίου Ροσφόρ ως προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 13. Πέρας. Εγκρίνεται. 17 για την, για την σκέψη Β. Εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 19 Μάντερς υπέρ κατά απορρίπτεται. 30 του κυρίου Ντεγιόγκ. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 30. Πέρας. Απορρίπτεται. 32. Άρχιδη ψηφοφορία για την 32. Πέρας. Εγκρίνεται. 35. Α, όχι. Πάμε στη συμβαστική 3 κατευθείαν. Uh, 3. Those Συμβιβαστική 3. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Περνάμε στη 46 τώρα, Μάγερ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Πηγαίνουμε συμβιβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στην 57. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στην 63. Σενάλοβα. Ποιοι είναι υπέρ. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 63. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 64. Χουάνγκ Νοκ. Ποιοι είναι υπέρ κατά, δεκτή. 65. Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. Κάποιο δεν ψήφισε. Όποιο δεν ψήφισε μπορούσε να αλλάξει το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία. Λοιπόν, να πατάτε τα κουμπάκια σα παρακαλώ. 66. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δύο εποχές, 16 υπέρ, 16 κατά απορρίπτεται. 68 ροσφόρ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 68. Τέλος. Δεκτή. 69. Ροσφόρ υπέρ. Κατά. Δεκτή. 67. Ντε Ιόγκ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ψηφίζουμε την 1. Τέλος. Απορρίπτεται. 2 και 3. Από κοινού ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτές. 4 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 5 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 6 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 7 υπέρ. Κατά. Τρελ Δεκτή. Περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Για το σύνολο του ψηφίσματος. Ψηφίζουμε. Ένας δεν έχει ψηφίσει ακόμα. Τέλος. Δεκτό το ψήφισμα. 30 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά και 2 αποχές. Η κυρία Χέντ ε, θα αλλάξει την ψήφο της. Ήθελε να ψηφίσει υπέρ. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε για μια ακόμη φορά για να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Το σύνολο του ψηφίσματος. Λοιπόν. Όσο περισσότεροι υπερψηφίσουν την έκθεση αυτή τόσο το καλύτερο. Τέλος. 30 υπέρ, μία ψήφος κατά και τρεις αποχές. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, συγχαίρουμε τον κύριο Κρόιτσμαν για μια πολύ δύσκολη έκθεση. Μετά από το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε, νομίζω ότι η έκθεση αυτή θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα υπάρξει και μια καλή συζήτηση στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν, ιδιαίτερα τους σκιώδεις εισηγητές. Κύριε Κρόιτσμαν, θέλετε να πείτε κάτι για να κλείσετε. Ευχαριστώ όλους. Ε, ο στόχο του εισηγητή είναι πάντα να έχει μεγάλη πλειοψηφία, γιατί στην πράσινη βίβλο ήταν όλα ανοιχτά. Η Κομισιόν έλεγε δεν θέλει να κάνει κάτι, με ήθελε μετά κάτι ήθελε να κάνει. Ήταν λίγο ασαφή τα πράγματα. Τώρα λοιπόν έχουμε έτσι μια μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο, οπότε θα πιέσουμε την Κομισιόν να δράσει. Και η Κομισιόν γενικώ δεν είναι πολύ φίλο ε, των ε, των δράσεων, αλλά νομίζω ότι τελικά μόνο μέσω ε, επικουρικότητας μπορεί να γίνει να, προωθήσει, να προωθηθεί το θέμα αυτό. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε την ε, πλειοψηφία που έχουμε, έτσι ώστε η Κομισιόν να μπορέσει να έχει και ενισχυμένη συνεργασία και να προωθήσει και την ενισχυμένη συνεργασία μέσω των κρατών μελών. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει πια η Κομισιόν. Εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έχουμε αυτή την ε, πλειοψηφία και χαίρομαι που η Κομισιόν επιτέλους θα μπορέσει να κάνει κάτι. Ευχαριστώ όλους για την ψήφα σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Κρότσμαν, ο οποίος ήταν τόσο ανοιχτός στις συζητήσεις που είχαμε για την έκθεσή του. Όμως πρέπει να σας πω κάτι, ότι κάποιες από τις τροπολογίες που δεν καλύπτονταν από τις συμβαστικές, δεν ήμασταν υπέρ και συμφωνήσαμε για το περιεχόμενο ότι ίσως σε κάποια σημεία να ζητήσουμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Γενικά με την έκθεση συμφωνούμε, αλλά σας ε, λέω ότι υπάρχει η πιθανότητα να ζητήσουμε κάποιες κατατμήματα ψηφοφορίας. Σα το λέω μετά από το αποτέλεσμα αυτό της ψηφοφορίας που είχαμε. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. όταν το συζητήσετε στην πολιτική σας ομάδα, ίσως να υπάρξουν και άλλες τροπολογίες. Αυτή είναι η πολιτική, τι να κάνουμε. Κάποιοι ξέρουν περισσότερα, κάποιοι ξέρουν λιγότερα. Σίγουρα πάντως θα στηρίξετε την θέση της Επιτροπής μας. Δεν έχω αμφιβολία. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση που έχει να κάνει με τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Κύριε Λεγκρίπ, το κύριε Λεγκρίπ, πριν ψηφίσουμε, θέλετε να πείτε κάτι. Ξέρω ότι έχετε προσπαθήσει να πετύχετε συμβαστικές και εγώ είμαι σκιώδη. Οπότε, ξεκινάμε. Αμέσω συμβαστική τροπολογία αριθμό ανεπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οπότε τώρα περνάμε και πάμε στην τροπολογία αριθμό 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Για το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Τροπολογία 6. Ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία αριθμό 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 τώρα, πριν τριγάσει. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 18. Εδώ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία αριθμός 3 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Οπότε πάμε τώρα στην τροπολογία 26 του κύριου Σφαμπ. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται σαφώς. Τροπολογία 5, συμβαστική 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 33 τώρα της ηγήτριας υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 37, Λεκεγκάρτ ως προσθήκη υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 37 Λέκεγαρ, όχι αυτή καταπίπτει. 34. 34. 34 της κυρίας Πρέντεγαρτ. Υπέρ. υπάρχει κάποιο λάθος από ό,τι φαίνεται στον κατάλογο ψηφοφορίας. Γι' αυτό με την 37. Πάμε πίσω γιατί υπάρχει κάποιο λάθος. 33, εντάξει, πέρασε. 37, Λέκεγαρτ, απορρίφθηκε. 34 τώρα. Συμφωνεί η κυρία. Πριν κάνετε λοιπόν, 34. 34. Στην παράγραφο 5α νέα, έτσι, 34. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35 τώρα, του κύριο Καφά. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Πρέντε γάστ. Ψηφίστε παρακαλώ για την 39. Πολύ αργά πάει. Εντάξει, περιμένουμε ακόμα. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Εγκρίθηκε της κυρίας Πέντεκας. Ναι. Τελική γνωμοδότηση. Ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 32 ψήφοι υπέρ και δύο αποχές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λεγκρίπ. So I'm sure you will defend our opinion. Ε, θα πάτε και στην Διεθνή Επιτροπή έτσι και θα στηρίξετε τι δικές μας τροπολογίες. Τώρα, τελική ψηφοφορία, τελευταία ψηφοφορία είναι το σχέδιο γνωμοδότηση για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ιδίε πρωτοβουλία εκθεσή του για μια ε, συνεπή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις συλλογικέ προσφυγέ. Κύριε Ράπτη, θέλετε να πείτε δύο λόγια πρώτα, παρακαλώ. I to thank you all. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Με την υπόθεση αυτή ε, προχωράμε στις συλλογικέ προσφυγές. Συλλογική ένομη προστασία. Συνεχίζω στα ελληνικά, λέει η Μαλήτρια. Ε, δύο σημεία τα οποία θα ήθελα να πω πριν από τις ψηφοφορίες. Το ένα είναι καθαρά διαδικαστικό ε, κάναμε μία μικρή αλλαγή στην συμβιβαστική τροπολογία 8 επί της παραγράφου 12α, μία αλλαγή που έγινε δεκτή από όλες τις πολιτικές ομάδες και τις ευχαριστώ γι' αυτό. Και ακριβώς η αλλαγή αυτή αφορά την μεγαλύτερη ενημέρωση για την έναρξη μιας συλλογικής προσφυγής. Προτείνω για λόγους συνοχής του κειμένου μετά την υιοθέτηση της γνωμοδότησης και των τροπολογιών, αφού τελειώσουμε με την ψηφοφορία, να μετακινήσουμε την παράγραφο 16 μετά τη νέα παράγραφο 12α. Αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τις ε, ψηφοφορίες. Το δεύτερο ζήτημα είναι κάτι που λιγάκι με έχει στεναχωρέσει. Ε, έχει ζητηθεί ε, split vote και το split vote αυτό έχει ζητηθεί στη συμβιβαστική 5. Οι ομάδες ALDE, APP και ECR έχουν ζητήσει και οι πράσινοι έχουν ζητήσει αυτό το split vote. Ε, θέλω πριν ψηφίσουμε να πω δύο σκέψεις. Ε, τι αφορά το split vote. Το split vote αφορά το να μην περιλαμβάνονται οι λέξεις και για τις εθνικές υποθέσεις. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να περιλαμβάνονται αυτές οι λέξεις και national cases. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι αν οι δύο λέξεις βγουν, τότε αφήνουμε εκτεθειμένες στον αθέμητο ανταγωνισμό τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σωστά στις υπόλοιπες χώρες που δεν έχουν συλλογικές προσφογές. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ πως εάν φύγουν οι λέξεις national cases, ουσιαστικά αφήνουμε χώρο για το forum shopping. Και το forum shopping έχουμε πει ότι δεν το θέλουμε. Ε, το τρίτο και τελευταίο είναι ότι όλοι έχουμε τις πληροφορίες μας και ξέρουμε ότι η διαβούλευση που έχει γίνει ε, δείχνει ότι υπάρχει ε, πολύ μεγάλη θέληση των πολιτών της Ευρώπης για νομοθετική δράση τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο. Και σκέφτομαι, εμείς που είμαστε οι εκπρόσωποι των πολιτών, έχουμε το δικαίωμα να πάμε ένα βήμα πίσω από αυτό που θέλουν οι πολίτες. Έτσι, ε, ήθελα να ακούσετε αυτές μου τις σκέψεις ε, για το split vote που έχει ζητηθεί ε, στο Compromise 5. Ε, ε, κάτι τελευταίο και κλείνω είναι ότι είμαι σαφώς υπέρ της επικουρικότητας, είμαι σαφώς υπέρ των κοινών αρχών και σε καμία περίπτωση δεν μου αρέσει η επιβολή στα κράτη-μέλη. Με ενδιαφέρει η καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Εδώ κλείνω, βάζω μια τελεία και σας ευχαριστώ ξανά όλους. Okay. All right. Well, thank you for... Ωραία. Ευχαριστούμε. Θα τα ξαναδούμε και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ώστε να είναι σαφή τα πράγματα. Κύριε Σβάμπ, θέλετε να σχολιάσετε. Δεν θέλω να συζητήσουμε τώρα το θέμα. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Σύντομα. Θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ τη συνάδελφο αυτή για την εξαιρετική τη δουλειά και θέλω να πω ότι αυτή την τροπολογία για την ξεχωριστή ψηφοφορία που ζητήσαμε δεν την θέσαμε για να δημιουργήσουμε προβλήματα, αλλά γιατί ο σκιώδης εισηγητής μας, δυστυχώ δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ, μας ε, είπε για την νομική βάση για την παρέμβαση στην εθνική κυριαρχία για το σημείο αυτό, ότι είχε κάποιες αμφιβολίες. Βεβαίως είμαστε ανοιχτοί για τη, συζήτηση, αλλά δυστυχώς θέλουμε να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία, ε, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και τις φιλικέ σας ε, συμβούλες. Ευχαριστώ. Right, let's vote then. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ξεκινάμε με την τροπολογία 25. Κρόιτσμαν και Φόξ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία ε, συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 2. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 39. Φόξ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 37. Κρότσμαν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 40 καταπίπτει. Παράγραφος 5α, καινούρια. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική 5. Με ψηφοφορία κατά τμήματα που έχει ζητήσει το Άλντε και το ΕΛΚ. Το πρώτο τμήμα. Όλο το κείμενο χωρίς τις λέξεις both national and. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας 5. Πέρας. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Όλες οι υπόλοιπες τροπολογίες καταπίπτουν και πάμε στην στη συμβαστικη 5 5α. Συμβαστική τροπολογία 5α. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 62 της εισηγήτριας. Άρχεται η ψηφοφορία για την 62. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στην συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 66. 66. Άρχεται η ψηφοφορία για την 66. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στην 69 της εισηγήτριας με ψηφοφορία κατά τμήματα. Βλέπετε ποια είναι τα τμήματα, δεν χρειάζεται να σας το διαβάσω, τα βλέπετε στην, ε, στη λίστα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10. Τροπολογία 70. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 71. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 73. 73 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική 8. Πάλι ψηφοφορία κατά τμήματα. Βλέπετε ποια είναι το πρώτο και το δεύτερο κείμενο. Θα δίνονται σχετικές πληροφορίες σε όλου τους πιθανού καταναλωτέ. Το πρώτο τμήμα, χωρί αυτέ τι λέξει λοιπόν ψηφίζουμε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για το τμήμα 2. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 91 του κυρίου Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ετροπολογία 92 προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 95. 95 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική 10. Είναι 94 και 96 καταπίπτουν. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 103 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Α, συγγνώμη, έχει ψηφοφορία κατά τμήματα. Τώρα το είδα. Ωραία. Λοιπόν, συμβαστική 13, τμήμα 1. Υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 121 του κυρίου Χουάνγκ Νόκ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 121. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στην 122 της κυρίας Γκάλο. Ε, ψηφοφορία κατά τμήματα από το ΕΛΚ ζητήθηκε. Τμήμα 1. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για το τμήμα 1. Πέρας. Απορρίπτεται 16-16. Και το τμήμα 2 απορρίπτεται. Εκτιμώντας. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 30 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 1 αποχή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ όλους. Κυρία Ράπτη, θέλετε κάτι να πείτε, παρακαλώ. Άφησα για το τέλος τις θερμές ευχαριστίες στα γραφεία των σκιωδών εισηγητών και στη γραμματεία της Επιτροπής. Η βοήθειά τους ήταν πολύτιμη και νομίζω ότι πρέπει όλοι να τους ευχαριστήσουμε. Uh, Ωραία. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε τη συνεδρίαση για σήμερα. Στι 11 θα ξεκινήσει τη συνεδρίαση οι συγητέ, οι ε, συντονιστέ, συγγνώμη. Η επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στι 3 το απόγευμα. Θα σας δω τότε. Ευχαριστώ όλους όσους δεν θα παραμείνουν για την συνάντηση των συντονιστών.